αν δεν έχετε ε, παρατηρήσεις ε, θα την εγκρίνουμε και θα περάσουμε στο σημείο 3 κατευθείαν χωρίς να περάσουμε από το σημείο 2. Στη σύνδεση μέσω Skype με τον Joshua Wong, Γενικό Γραμματέα ε, του κόμματος Δεμοσίστο του Hong Kong ο κ. Κόφερ, πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τη σχέση με την Κίνα, βρίσκεται παρόν εδώ και είναι χρήσιμο να το κάνουμε συνήθεια. Να το κάνουμε σύστημα, να προσκαλούμε δηλαδή προέδρους αντιπροσωπιών όταν συζητούμε θέματα που έχουν σχέση με τις δικές τους αρμοδιότητες. Με αυτόν τον ε, τρόπο μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας ε, παρακολουθεί τα γεγονότα στο Χονγκ Κονγκ με πολύ ενδιαφέρον. Η κατάσταση του Χονγκ Κονγκ ήδη έδωσε θέση σε ένα ψήφισμα τον Ιούλιο. Το Σεπτέμβρη θελήσαμε να προσκαλέσουμε τον κύριο Τζόσουα Wong να έρθει σε, να μας δει προσώπο. Δεν έγινε αυτό, δεν κατέστη δυνατό, αλλά σήμερα είναι μαζί μας, έστω και μέσω Skype. Καλημέρα Τζόσουα Wong. οι νέες τεχνολογίες πραγματικά τίθενται στην υπηρεσία της ελευθερίας έκφρασης αλλά μερικέ ε, φορέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να περιοριστεί η ελευθερία έκφραση. Αυτό το βλέπουμε σε ορισμένε χώρε και βέβαια ιδιαίτερω στην Κίνα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπιουτικόφερ, για μια σύντομη εισαγωγή. Να σας υπενθυμίσω ότι τα γεγονότα στο Χονγκ Κόνγκ ε, καθιστούν αυτή τη στιγμή ε, γίνονται αυτή τη στιγμή ε, το σημείο στο οποίο είναι πιο έντονη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Είμαστε σε επαφή με τους διαμαρτυρόμενους στο Χονγκ Κόνγκ και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε ως αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Κίνα. Να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των ε, τελευταί, τελευταίων εκλογών για τα διαμερισματικά διαμερισματιακά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια στο Χονγκ Κόνγκ δημιούργησε ε, μια καινούργια κατάσταση. Ε, ήταν συντριπτική η νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων. Πιο εντυπωσιακή από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στην πρόσφατη ιστορία. Αυτό αποδεικνύει κάτι το οποίο κάποιες πλευρές αμφισβητούσαν. Ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ στηρίζουν ε, και βρίσκονται στο πλευρό του δημοκρατικού κινήματος. Σε, αυτή την, σε αυτό το καινούριο πανόραμα θα ήταν καλό Οι κυβερνητικές αρχές του Χονγκ Κονγκ και οι ηγέτες τους στο Πεκίνο να προβληματιστούν και να ακούσουν την φωνή των πολιτών του Χονγκ Κονγκ. Ε, δύο είναι τα αιτήματα των πολιτών, τα βασικά τους αιτήματα, τα οποία υποστηρίζει σίγουρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του ψηφίσματος στο οποίο, ανέφερε, στο οποίο αναφέρθηκε η Πρόεδρος. Πρώτον, μια ανεξάρτητη έρευνα για, τις, για τη βάναυση συμπεριφορά της αστυνομίας και δεύτερον, μια καινούρια ε, εκκίνηση, μια καινούργια αφετηρία για την καθολική ψηφοφορία στο Χονγκ Κονγκ. Η Κάρι Λάμ, η του εκτελεστικού στο Χονγκ Κονγκ και το Πεκίνο μέχρι τώρα δεν έχουν ε, ε, εισακούσει τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ, αλλά εμείς θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι τους στηρίζουμε, είναι πάγια η θέση μας αυτή και ότι επιθυμούμε μια ειρηνική ε, ε, επίλυση του ζητήματος σύμφωνα με, τις, τα αιτήματα των δημοκρατικών του Χονγκ Κονγκ. Τζόσουα, έχεις το λόγο. So, you have the floor. For 10 minutes. Για 10 λεπτά. Okay, thank you. Thank you. Okay. Good afternoon. May I first... Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να εκφράσω την αγνωμοσύνη μου για την ευγενική σας πρόσκληση για να σας ε, αναφέρω το τι γίνεται στην ε, χώρα μου παρά τις, ε, τους περιορισμούς. Όταν μου απέρριψαν την αίτηση να ταξιδέψω, αισθάνθηκα πολύ χειρότερα από το να μου έβαζαν να, να με φυλάκιζαν. Γιατί δεν θα μπορούσα να έρθω στην, ε, στις Βρυξέλλες και να σας μιλήσω για τον αγώνα που κάνουμε για δημοκρατία και ελευθερία. Ξέρετε ότι ε, έγινε, υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή στις τελευταίες ε, εκλογές. Είχαμε 3 εκατομμύρια συμμετέχοντες, ψηφίσαντες. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνη προς τις αρχές του Πεκίνου η συμμετοχή έφτασε το 85% στην ε, χώρα και πάρα πολλές θέσεις ε, που μέχρι τώρα ε, τηρούνταν από κυβερνητικούς συνασπισμούς τώρα έχουν αναλυφθεί από τους διαδηλωτές, από τους ανθρώπους που μπορούν να εξασφαλίσουν δημοκρατία, ελεύθερες εκλογές. Το Hong Kong βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση η οποία πρέπει να λυθεί με πολιτικό τρόπο, αντί για καταστολή από την αστυνομία. Αυτά είναι τα αιτήματα, τα οποία όμως μας αρνούνται να μας αναγνωρίσουν. Υπάρχει μεγάλη καταπάτηση των πολιτικών ελευθεριών στην αρχή διαδηλώναμε The government arrest me and charge me of decided people taking part in an unauthorized assembly. Then I went contesting in this local election on Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα στον ήχο και η διερμηνία δεν μπορεί να συνεχίσει. Political censorship.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 I was arrested for three times, prosecuted, and later imprisoned for my leading role in the umbrella movement. My colleague Nathan Law, the youngest lawmaker in... Ο συνάδελφός μου επίσης συνελήφθη και ε, φυλακίστηκε. Έχουμε κατανοήσει ότι υπάρχει σημαντική καταστολή. Κινέζικα στρατεύματα αναπτύχθηκαν το Χονγκ Κονγκ, στρατιώτες στο γύρω-γύρω από, το, ε, από την Πολυτεχνιούπολη, έκλεισαν τους δρόμους, Αυτή είναι πραγματικά η επιθετική συμπεριφορά της ε, Κίνας και πρέπει να υπάρξει παγκόσμια αντίδραση. Τους τελευταίους μήνες Μιλώ με πολλού δημοσιογραφού από όλο τον κόσμο που θέλουν να αναφέρουν το τι γίνεται στο Χονγκ Κονγκ και θα ήθελα και να στείλω σε εσά ένα μήνυμα. Καταρχάς η αστυνομική βία είναι πολύ πιο σοβαρή από αυτά που αναφέρουν τα μέσα. Υπάρχουν ξυλοδαρμοί από τους αστυνομικού, υπάρχουν βιασμοί εντό των αστυνομικών τμήματων και επίσης υπάρχουν, υπάρχει ε, καταστολή σε ό,τι αφορά τις ε, ε, εκτρώσεις. Θέλω λοιπόν να μιλήσω στην διεθνή κοινότητα να σταματήσει αυτή την ανθρωπιστική κρίση για να μην βαρυνθεί περισσότερη κατάσταση. Επίσης, πρέπει να υπάρξει, υπάρχει μάλλον μετα, ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των διαδηλωτών. Οι εκλογές και το διεθνές lobbying είναι παραγωγέ που μπορούν να βοηθήσουν το κίνημά μας για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ελευθερία μετακίνηση. Θέλουμε να έχουμε ελεύθερες εκλογές και κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη νίκη, αλλά έχουμε, κάνει, έχουμε πετύχει κάποιες μικρές νίκες. Είναι Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για να υπάρξει όντως εγκαθίδρυση της ε, δημοκρατίας μετά από λαϊκή εντολή. Είναι ηρωνικό το ότι το Χονγκ δεν μπορεί να έχει ελεύθερες εκλογές ε, λόγω της ε, απολυταρχίας του Πρόεδρου Σι. Από τον Ιούνιο φέτος οι διαδηλωτές ε, αντιμετωπίζουν χτυπήματα από σφαίρες. Υπάρχουν μάλιστα ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δίνουν ε, ε, ε όπλα σε αυτούς τους ε, για να καταστήλουν το κίνημα. Το Χονγκ Κόνγκ είναι πραγματικά ιστορική πόλη δεν ξέραμε ποια είναι η, η πρόθεση του, του κινέζικου καθεστώτος να παρακολουθεί την οικονομία και τη ζωή μας στο Χονγκ Κόνγκ. Η οικονομία μας αυτή τη στιγμή επαφίεται στην κατάσταση στην Κίνα και γι' αυτό, αυτό κάνει πιο ε, δύσκολη την, τον αγώνα μας για ελευθερία. Πρέπει να σταματήσουμε να ε, επαφιέμεθα και να εξαρτώμεθα από την οικονομική κατάσταση στην Κίνα. Πολλοί θα πούν ότι ανησυχώ πάρα πολύ ή κατακρίνω πολύ την Κίνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Κίνα δεν παίζει με τους, σύμφωνα με τους κανόνες. Έχει πραγματικά α, δεινό παρελθόν στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν τιμά τις διεθνείς συνθήκες και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι οι οποίοι ε, βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε στρατόπεδα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και βρίσκονται σαν φυλακισμένοι. Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται. Γι' αυτό εγώ κάνω έκκληση σε πολιτικούς και ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να είναι στο πλευρό των διαδελωτών στο Χονγκ Κονγκ που παλεύουν για έναν πραγματικά α, σημαντικό στόχο αυτών των ελεύθερων εκλογών. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ξανασκεφθούν τις, ευρωπα... τις οικονομικές σχέσεις που έχουν με αυτό το πολιταρχικό καθεστώς που δεν παίζει ποτέ με τους κανόνες. Υπάρχει υπάρχουν διάφορες διεθνείς πράξεις οι οποίες θα πρέπει να τιμηθούν για να σταματήσουν υπεραιτέρω παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Χονγκ αλλά και σε άλλα σημεία της Κίνας. Τέλος, καταλαβαίνω ότι οι επιχειρηματίε και οι πολιτικοί ανησυχούν ότι αν, αν σταθούν απέναντι στην Κίνα για, την, για τις καταπατήσεις των δικαιωμάτων μπορεί να επιβαρύνει αυτό, να επιδεινώσει τις σχέσεις τους. Αλλά θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να είναι και αληθινές στις αξίες που, α, στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ούτε έμεσα ούτε άμεσα να ε, ενθαρρύνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο υπόλοιπο ελεύθερος κόσμος θα πρέπει να σταματήσει να κάνει ότι δεν βλέπει. Η θέση μας είναι σαφής. Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ υπερασπίζονται όχι μόνο τις ατομικές πολιτικές ελευθερίες, αλλά και τις δημοκρατικές αξίες, την οικονομική ελευθερία σε αυτή την διεθνή πόλη. Είμαστε απέναντι στο πολιταρχικό καθεστώς και θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για δημοκρατία. Γιατί δεν θέλουμε ούτε πολιτερχικό κράτος να γίνουμε, ούτε αστυνομικό. Με είμαι ο Τζόσουα Γουόν και έχω συλληφθεί από την αστυνομία, αλλά θα συνεχίσω να παλεύω για, στο πλευρό των διαδηλωτών για να έχουμε τελικώς ελεύθερες εκλογές και να εκλέξουμε την κυβέρνησή μας. Κάνω έκκληση λοιπόν σε εσά να σταθείτε στο πλευρό των πολιτών του Χονγκ Κόνγκ. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζόσουα. Ευχαριστώ που αναφέρθηκε στο άρθρο 21 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, ε, συνθήκης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ για τον αγώνα που δίνεται στο Χονγκ Κονγκ. Θα δώσω το λόγο στα μέλη που είναι παρόντα. Ποιος θα ήθελε να μιλήσει, Ισαβέρα Βίσλε. Ευχαριστούμε πολύ για τις δηλώσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό για μας που έχουμε την άμεση αυτή επαφή μαζί σας. Σας θαυμάζουμε για το κουράγιο σας, το δικό σας και αυτόν που αγωνίζονται μαζί σας. Μα είμαστε πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα των εκλογών εδώ στην Ευρώπη είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση, ποια είναι η δική σας εκτίμηση μπορεί να είναι μήνυμα αλλαγή το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Μετά, ποια είναι τα επόμενα βήματα Ποια είναι τα βήματα τα οποία θα αναλάβετε εσείς και τι είναι δυνατόν να κάνετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Επίσης, ποια είναι τα βήματα τα οποία περιμένετε από την κυβέρνηση και πώς μπορούν τα αποτέλεσμα των εκλογών, των πρόσφατων εκλογών, να επηρεάσουν την κυβέρνηση. Τέλος, η ερώτηση που πάντοτε θέτουμε, ε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να σας βοηθήσουμε. Προφανώς σας δίνουμε το λόγο, μας μιλάτε, είναι μια πρώτη βοήθεια. Τι άλλο όμως μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. I give the floor to for the... Ο κ. Γκλουξμαν για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσία σας έστω και μέσω Skype. Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να σας έχουμε αυτοπροσώπως. Είναι κρίμα ε, που έχει ληφθεί η απόφαση απαγόρευση ταξιδιού. Ευχαριστούμε πολύ για τον αγώνα σας. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το κίνημά σας. Και ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε και στα άλλα θύματα ε, του, των γενεζικών πράξεων, τους Ουιγούρους για παράδειγμα. Ε, πολύ μεγα, ένα πολύ μεγάλος αριθμός σιγουρών βρίσκονται σε στρατόπεδα κράτηση, Και εγώ ήθελα να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και πιο συγκεκριμένα αναφερθήκατε στις ευρωπαϊκές εταιρείε, οι οποίες πολλούν εξοπλισμό ε, στις κοινωνικές αρχές, ε, εξοπλισμός ο οποίος χρησιμεύει αργότερα στις αστυνομικές αρχές Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Αν αποδειχθεί ότι ε, ευρωπαϊκές εταιρείες βοηθούν ε, τις κινέζικες αστυνομικές αρχές ε, να συντρίψουν το κίνημά σας, μπορούμε να λάβουμε μέτρα. Ευχαριστώ. Η Ειρήνα Φομβέση. Thank you very much, Mr. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Wong Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία και έτσι μπορούμε να σας δούμε και να σας ακούσουμε παρά την ταξιδιωτική απαγόρευση. Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Μου φαίνεται, και δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε, ότι οι κινέζικες αρχές έχουν βρει ένα νέο όπλο, την παραπληροφόρηση. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές αντικρουόμενες εκθέσεις ε, στα μίντια και είδα ότι και η Ρωσία παίρνει το μέρος της Κίνας και ότι ήταν ιδιαίτερα αρνητική όσον αφορά τις διαδηλώσεις. Και προβλήθηκε ιδιαίτερα η βία εκ μέρους των διαδηλωτών. Ξέρουμε ότι υπήρχαν προβλήματα με κάποιους προβοκάτορες. Είναι λοιπόν αυτό το νέο όπλο της Κίνας, η παραπληροφόρηση. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, για να την αντικρούσουμε. Και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, για να μπορέσουν να συμμετέχουν οι χώρες της Ένωσης και να παραμείνουν ειρηνικές οι διαδηλώσεις, είναι ακριβώς λοιπόν αυτό. Και όσον αφορά τον νόμο που πέρασε την περασμένη εβδομάδα, που πέρασαν οι ΙΠΑ για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, ποια θα είναι η ε, επιρροή του. Μα είπατε ότι ίσω και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα υιοθετώντα μια ανάλογη νομοθετική πράξη. Julie έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τζόσουα, χαίρομαι Ιδιαίτερα που είσαι μαζί μας σήμερα, αλλά λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να σε συναντήσω αύριο όπως είχαμε προγραμματίσει. Είμαι Βρετανή και έχω συνεργαστεί με τους Βρετανούς σοσιαλιστές που στηρίζουν το κίνημά σας. Και βεβαίως ε, υπήρχε και το θέμα με την Κατάι Πασίφικα. Κάναμε λοιπόν ε, μία αναφορά το καλοκαίρι με περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Ελπίζω ότι μπόρεσες να δεις αυτή την αναφορά ε, εδώ στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Είναι ένα βρετανικό πρόβλημα, αλλά όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικές σχέσεις με άλλες χώρες, είναι γνωστό. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς μπορείς εσύ να μας βοηθήσεις, διότι εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο η δεξιά και η αντιευρωπαϊκή ε, αυτοί που είναι κατά της Ευρώπης υποσκάπτουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τη στήριξή σου προκειμένου να καταρρύψουμε κάποια από τα επιχειρήματά τους. Σα ακούω να μας μιλάς ανοιχτά και εκτιμάς ιδιαίτερα αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, να τα προωθήσουμε, να αντισταθούμε σε καταχρήσεις ε, ε, ισχύω. Έχουμε όμως και εμείς τις δικές μας μάχες εδώ. Και πρέπει να πω ότι το Hong ε, στην Ολομέλεια συζητήθηκε ιδιαίτερα και χρησιμοποιήθηκε. και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη στήριξή σου, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της υπόσκαψης της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Μπέχναρ Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα είναι στο Χονγκ Κόνγκ. Μια πολύ απλή ερώτηση. Υπάρχει κάποιο στο Χονγκ Κόνγκ άντρα ή γυναίκα που θα μπορούσε να κάνει τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στο δημοκρατικό κίνημα και τις αρχές του Πεκίνου για να διαπραγματευτεί κατά κάποιον τρόπο, ε, να μπορέσει να βρεθεί έτσι μια πολιτική ένας πολιτικός συμβιβασμός. Τζόσουα, έχει τον λόγο για να απαντήσει αυτέ τι ε, ερωτήσει και ίσω στη συνέχεια κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Αλλά στην αρχή απαντά αυτέ τι ερωτήσει, έχει τον λόγο. Για το αποτέλεσμα των εκλογών, 70% των ψηφισάντων ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή με πάνω από 85 100 ε, των ε, συμβουλίων έχουν κερδιθεί από ε, φιλοδημοκρατικέ δυνάμει. Φαίνεται λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η νίκη και φαίνεται πόσο πολύ δεν εμπιστεύονται οι πολίτε στο Πεκίνο. και φαίνεται ότι είναι και μεγάλη η στήριξη προ του διαδηλωτέ. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό μήνυμα για την καταστολή που δείχνει η κινέζικη κυβέρνηση. Ο μόνο τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα είναι να υπάρξουν συμβιβασμοί και διαπραγματεύσει με του πολίτε του Χονγκ Κόνγκ. Τώρα για την καταστολή των διαδηλώσεων, πάνω από 5.800 άνθρωποι συνελήφθησαν, τουλάχιστον 500 εκ των οποίων ε, αντιμετώπισαν διώξεις, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μπορεί να μπουν στη φυλακή για 10 χρόνια. Λίγα, λίγους μήνες πριν, το καλοκαίρι, οι αστυνομικές δυνάμεις συνελάμβαναν ακτιβιστές από το Σεπτέμβρη και μετά ή τον Οκτώβρη είναι πολύ αυθαίρετο ο τρόπος που συλλαμβάνουν πολίτες. Όχι μόνο διαδηλωτές ή ακτιβιστε συλλαμβάνουν και θρησκευτικού θρησκευτικούς γιατρού, γιατρούς, ε, νοσοκόμους, άτομα που δίνουν πρώτες βοήθειες. Επίσης συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Γι' αυτό μιλώ για ανθρωπιστική κρίση. Ακόμα και κατά τη διάρκεια πολέμου, ο στρατό δεν συλλαμβάνει νοσοκόμου και γιατρού. Τώρα, για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε πώς το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχει συμφωνήσει να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων προς τις αστυνομικέ δυνάμεις του Χονγκ Κονγκ. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα ε, υιοθέτησε νομοθεσία για να στείλει σαφή, σαφές μήνυμα για το πώς η, Ευρωπα... δεν θα στείλουν εξοπλισμό ή οπλισμό στις ε, δυνάμεις του Χονγκ Κονγκ. Ε, είχαμε ας πούμε ε, εκτοξευθύρες νερού. Ε, οχήματα για, να, για τη διαχείριση των πληθών είχαν επίσης εξαχθεί από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Οπότε νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτές οι χώρες πρέπει να σταματήσουν τις εξαγωγές. Λίγες μέρες πριν, ο αρχηγός, ο διευθυντής της ε, αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ τόνισε το ότι αν δεν μπορούν να υπάρξουν, αν δεν μπορούν να υπάρξουν εξαγωγές από, την ΙΠΑ, από τις ΗΠΑ ε, όπλων ε, και εξοπλισμού θα, θα προσπαθήσουν να τις πάρουν από την Ανατολική Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταθούν στο πλάι του Χονγκ Κονγκ. Τώρα, για το θέμα των διαπραγματεύσεων. Οι φιλοδημοκρατικοί ηγέτες προσπαθούν να κάνουν διαπραγματεύσεις ήδη από τον ε, Ιούνιο με την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, αλλά η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ δεν λαμβάνει αποφάσεις. Δεν είναι ε, κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τους πολίτες. Παίρνουν διαταγές από το Πεκίνο είναι πιστή στο Πεκίνο. Ακόμα και ο διάλογος να γίνει με την κυβέρνηση, ε, με αξιωματούχους της κυβέρνησης, δεν θα γίνει, δεν θα είναι αποτελεσματικό, γιατί απλώς κάνουν ότι δεν βλέπουν και συνεχίζουν την καταστολή των διαδηλώσεων. Παρόλο που είχαμε τεράστια επιτυχία στις εκλογές η αστυνομία εξακολουθεί να πυροβολεί με πλαστικές σφαίρες σε μεγάλες εμπορικές περιοχές του Χονγκ Κονγκ. Για να κλείσω λοιπόν, στηρίξτε το Χονγκ Κονγκ, εσείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι θέμα ε, ε, ε, είναι θέμα του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. έχουμε σταθεί απέναντι στην καταστολή από την κυβέρνηση σε αυτή την παγκόσμια πόλη. Η πράξη για τη δημοκρατία θα πρέπει να τύχει σεβασμού. Και καλό θα ήταν ίσως να έχουμε και κάποιους μηχανισμούς ε, κυρώσεων για να, με στόχο τους αστυνομικούς, ε, τις αστυνομικές ε, δυνάμεις ή τους πολιτικούς. Ελπίζω οι απαντήσεις μου να σας διαφωτίζουν λίγο και να ρίχνουν λίγο φως στην κατάσταση για το ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, σίγουρα ένα από τα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι η ε, πάυση των εξαγωγών. Εμείς θέλουμε στήριξη από εσά αλλά και από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα. Είπες ότι η οικονομία του Χονγκ Κόνγκ σχετίζεται με την οικονομία του Πεκίνου και αυτό είναι απειλή για το Χονγκ Κόνγκ. Είναι πλεονέκτημα όμως να είναι κανείς το οικονομικό κέντρο όπως είναι το Χονγκ Κόνγκ και το Πεκίνο. Και εμείς έχουμε κάποια σχέση με αυτό, γιατί ξέρετε ότι πολλές επενδύσεις έρχονται από την Ευρώπη προς το Πεκίνο και οι επενδύσεις αυτές γίνονται στο Χονγκ Κόνγκ. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα με κάποιο τρόπο. Το Χονγκ Κόνγκ είναι όντως ένα διεθνές οικονομικό κέντρο και έχει αναγνωριστεί ως τέτοιο. Είναι μια παγκόσμια οικονομική πόλη. Είναι σημαντικό το πλεονέκτημα που έχει το Χονγκ Κονγκ εδώ και δυο τρει δεκαετίες ή ίσως ε, και πιο νωρίς από τότε που γεννήθηκα εγώ. Τα τελευταία δέκα χρόνια, από τότε που ο Xi Jinping πήρε την ε, εξουσία και διοικεί, ήταν σημαντική η αλλαγή των ε, ντόπιων πλουσίων, οι οποίοι τώρα τη χάνουν εκμετάλλευση από τους επιχειρηματίες του Πεκίνου. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική ε, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από δύο δεκαετίες. Τώρα, πώς θα διατηρηθεί η οικονομική ελευθερία του Χονγκ Κόνγκ, αυτό είναι όντω πάρα πολύ σημαντικό. Οι ευρωπαϊκέ χώρε θεωρώ ότι πρέπει να κάνουν εμπορικές συμφωνίες με την με το Χονγκ αλλά μέσω μιας διαφορετικής πλατφόρμας, μέσω διαλόγου ή διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι σημαντικό όταν κάνουμε συζητήσεις για τις εμπορικές συμφωνίες και βεβαίως αναγνωρίζουμε και την ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν λέω ότι είναι ώρα να σταματήσουν όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί η πολιτική αστάθεια που υπάρχει και να υπάρξει πίεση στην κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, στην κυβέρνηση του Πεκίνου, για να τους θυμίσουμε ότι τώρα είναι ώρα να λυθεί το ανθρωπιστικό πρόβλημα, η ανθρωπιστική κρίση και να δούμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ. Να βάλουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ατζέντα. Αυτό νομίζω ότι είναι το, αυτό που περιμένουν τώρα οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ε, ε απάντησή σας. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θίξω τρία ζητήματα, Τζόσουα. Όταν ξεκίνησε την παρουσίασή σου αρχικά, μίλησες για μια πολιτική λύση. Επίσης είπες και τη λέξη συμβιβασμός, δύο φορές μάλιστα. Η ερώτησή μου είναι, μια πολιτική λύση που θα συμπεριλαμβάνει κάποιο συμβιβασμό. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς διαπραγμάτευση με τις αρχές του Χονγκ Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Οπότε, προκύπτει το εξή ερώτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συντροπτική στήριξη της ε, ε, του δημοκρατικού κινήματος από τους ε, πολίτες του Χονγκ Κόνγκ. Αυτό το γεγονός δεν μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα έτσι ώστε το δημοκρατικό κίνημα ε, να δείξει συμβιβαστικές διαθέσεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με εσάς να έχετε το πάνω χέρι. Επίσης, Είδαμε την Κυριακή πολλά επεισόδια στους δρόμους ε, και εσείς ε, ε, καταγγείλατε βία της αστυνομίας. Σωστό. Είδαμε όμως και άλλου τύπου βία. Μπορεί να ήταν προβοκάτος, μπορεί και όχι όμως. Αυτού του είδους η βία όμως δεν διευκολύνει την πρόθεση της δημοκρατίας. Και αυτό θα πρέπει να το καταστήσω σαφές. Τρίτον, το νόμο τον οποίο υπέγραψε πριν μερικές μέρες ο κύριος Τραμπ. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη ευρεία πλειοψηφία έχουμε ζητήσει ένα, να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Τα κράτη-μέλη όμως ε, δείχνουν επιφυλάξει προς το παρόν. Είναι φυσιολογικό παρόλα αυτά να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν όμως αρχίσουμε να στηρίζουμε ad hoc κυρώσει εναντίον της α της β χώρες χωρίς αυτές να εμπίπτουν σε ένα παγκόσμιο μηχανισμό θα ήταν σαν να υποσκάπτουμε τις προσπάθειές μας. Ασφαλώς και θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε το Χονγκ Kong ε, στο γενικότερο πακέτο αλλά δεν θα ήθελα να εγκαταλείψουμε την ε, σφαιρική μας προσέγγιση και να περάσουμε σε ad hoc κυρώσεις όπως εσύ ζήτησες. Η Λάουρα. Συνεχίζοντα την ερώτηση της κυρίας Αρένα, δεδομένου ότι το Χονγκ Κονγκ είναι οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο, υπάρχουν στο Χονγκ Κονγκ πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες και πολλοί ευρωπαίοι πολίτες που ζουν εκεί. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια και για αυτούς. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα θα έχουν μείνει στο περιθώριο των διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών. Είναι αλήθεια αυτό. Ε, πιστεύετε ότι έχουν να παίξουν κάποιο ρόλο οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις μας που βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ. Τέλος ο κύριος Γκέτα. Ε, ως συνέχεια της ερώτηση του κυρίου Μπιτουκόφερ. Δεν απαντήσατε στο ερώτημα μου για, για ένα ενδιάμεσο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο δημοκρατικό κίνημα στο Χονγκ και τις αρχές του Πεκίνου. Την ξεχάσατε την ερώτησή μου ή την αποφύγατε. Τζόσουα, έχεις το λόγο. Δυστυχώς και πάλι έχουμε προβλήματα με τον ήχο. Έχουμε συνεχείς διακοπές comment. You, you have to use your microphone because it's difficult to hear you. Yeah. Let me hold them. Thank you. Yeah. Thanks. Okay. Uh, first about. Αντί να καταδικάζουμε τους ίδιους τους ε, διαμαρτυρόμενους, ε, θα ήθελα να καταλάβουμε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι διαδηλώσεις. Ε, ε, η δική μας πρόσθεση ήταν να είμαστε να διαδηλώνουμε ειρηνικά αλλά δεν μας επιτρέπουν ελπίζω να το κατάλαβετε αυτό εγώ εξακολουθώ να πιστεύω στον ειρηνικό ακτιβισμό Ενδεχομένω δεν συμφωνώ με όλες τις πράξεις των διαδηλωτών, Όμω όπω είπα και προηγουμένω. οι, αυτοί που ασκούν βία μπορούν να διωχθούν, όμως η βία της αστυνομίας παραμένει ατιμόρυτη. Κανένας από τους αστυνομικούς δεν διώκεται για οτιδήποτε. Για παράδειγμα, για αυτά που συνέβησαν στο κάμπους, το πανεπιστημιακό κάμπους. Όταν ένα αστυνομικό όχημα ε, επιτέθηκε ε, σε φοιτητές όπως ακριβώς το τάξη Tiananmen Square στην πλατεία Tiananmen χρόνια πριν. δεν θα... Εμείς ζητούμε μια ειρηνική λύση προκειμένου να σταματήσει η βία και από τις δύο πλευρές προφανώς. Και, και εδώ περνάω στη δεύτερη λύση. Αν υπάρχει περίπτωση να γίνουν διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. για να αμβληθούν οι εντάσεις. Την 1η Ιουλίου, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να μπουν στο κοινοβούλιο, Ένας βουλευτής ζήτησε να ξεκινήσει διάλογος. Αργότερα η Κάρι Λαμ, η επικεφαλής ε, της ε, διοίκησης του εκτελεστικού, ε, διαφώνησε. Πολλοί όμως άλλοι βουλευτές και άλλοι άνθρωποι που στηρίζουν το Δημοκρατικό Κίνημα ζήτησαν αργότερα ε, διαπραγματεύσεις, αλλά και πάλι η Κάρι Λαμ τις απέρριψε. Οπότε, δεν έχουμε κανένα είδου επαφή αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κλείσει τα αυτιά και τα μάτια. Και αγνοεί τις, ε, τα αιτήματά μας. Τώρα, τι γίνεται με του επιχειρηματίε, του Ευρωπαίου επιχειρηματίε που βρίσκονται στο Χονγκ Κόνγκ και του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από τρει εβδομάδε, εργαζόμενοι ε, επιχειρήσεων ε, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Χονγκ Κόνγκ, πολύ κοντά στο χρηματιστήριο. Φορούσαν κοστούμια, ε, γραβάτες και ε, συναντήθηκαν ε, με το σύνθημα «Πολεμήστε για την ελευθερία σας» ε, ειρηνικά κατά τη διάρκεια του γεύματος, του μεσημερινού γεύματος. Διαλύθηκαν από την αστυνομία του Χονγκ Κόνγκ και κάποιοι μάλιστα συνέληφθησαν. Είναι, νομίζω, έχει έρθει η στιγμή, νομίζω, επιχειρηματίε και εργαζόμενοι από την Ευρώπη να ζητήσουν ε, μια, να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα για αυτά τα επεισόδια, όπως και για όλες τις βαρβαρότητες της αστυνομίας, οι οποίες μπορεί να συνεχιστούν και το 2020 παρόλες τις ελπίδες μας. Ε, η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ όμως ε, δεν δείχνει τάσεις να δώσει λόγο για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Φρόντισε τον εαυτό σου. Πρόσεξε και ελπίζουμε να σε δούμε εδώ στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Ε, είμαστε μαζί σας και σας υποστηρίζουμε. Συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν κατάφερα να έρθω αυτοπροσώπος. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή το δικαστήριο θα άρει την απαγόρευση ε, να εγκαταλείψω τη χώρα. Αλλά φαίνεται ότι ο περιορισμός της ελευθερίας ε, κίνησης ε, στο Χονγκ Κόνγκ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κίνας, της κυβέρνησης της ελπίζουμε και εμείς στο Χονγκ Κόνγκ όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ε, να μπορέσουμε να ασκήσουμε στο μέλλον τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Μπορείς να συνεχίσεις να μας ακούς γιατί θα μας ε, μιλήσει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε αν θέλεις μπορείς να συνεχίσεις στη σύνδεση. Και τώρα δίνω τον λόγο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Τζόναθαν Χάτουελ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε με πολύ σεβασμό και μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση του Joshua Wong και τις ερωτήσεις σας. Είχα πάει στο Χονγκ Κόνγκ την περασμένη εβδομάδα και ήμουν εκεί την Κυριακή των εκλογών. Ήταν μέρος μιας αποστολής που διεξήχθη εκεί Και πρέπει να πω ότι οι εκλογές ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστες, ήταν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα. Όχι μόνο διότι διεξήχθησαν ομαλά, γνωρίζοντας βέβαια τις πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά και γιατί έλαβαν χώρα με έναν τρόπο πολύ ειρηνικό, με πολύ σεβασμό. Κέρδισαν, όπως είπαμε, οι φιλοδημοκρατικές δυνάμεις και όπως είπε και ο Τζόσουα Βόγγ ήταν εμβληματικά τα αποτελέσματα. Διότι οι προδημοκρατικές δυνάμεις ε, κατέλαβαν τα 17 από τα 18 περιφερειακά συμβούλια. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα. Αυτό ήταν ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα εκ μέρους ε, του λαού του Χονγκ είναι κάτι που αμφισβητεί το αφήγημα που προωθεί τόσο η κυβέρνηση του Χονγκ όσο και η κυβέρνηση του Πεκίνου όταν λέει ότι ενεργεί εκ μέρους της σιωπηρής πλειοψηφίας. Το μήνυμα λοιπόν ήταν ξεκάθαρα υπέρ των δημοκρατικών δυνάμεων και της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ υπέρ των θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας. Η βία διεκόπη κατά τη διάρκεια των εκλογών, παραμένει ήρεμη κατάσταση και αυτό βεβαίως παρήχε μια ευκαιρία. Το Ευρωκοινοβούλιο, από τότε που κλιμακώθηκαν οι διαμαρτυρίες, από τον Ιούνιο δηλαδή, ε, έκανε διαρκή έκκληση για διάλογο για αποφυγή της κλιμάκωσης. Και πρόσφατα είχαμε την ε, ανακοίνωση της ύπατης εκπροσώπου που διασαφήνισε ότι οι διαμαρτυρίες ναι μπορεί να γίνονται ειρηνικά αλλά η χρήση βίας εκ μέρους της αστυνομίας η αντιμετώπιση ήταν πραγματικά δυσανάλογη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει έρευνα για την χρήση της βίας και τα αιτιά της. Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πώς οι αρχές του Χονγκ Κόνγκ θα αντιδράσουν σε αυτά τα ξεκάθαρα αποτελέσματα των εκλογών και κατά πόσον είναι έτοιμες οι αρχές αυτές να διαπραγματευτούν, ποια θα είναι η πολιτική ανταπόκριση. Είναι ξεκάθαρο βεβαίως ότι χρειάζεται, ναι, πολιτική ανταπόκριση, διαδικασία διαλόγου και ότι θα πρέπει αυτός ο διάλογος να ανήκει στο Χονγκ Κόνγκ. Όμως έχουμε και τη θέση του Πεκίνου που είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ. Οποιαδήποτε λύση στην κατάσταση για το Χονγκ Κόνγκ θα είναι αδύνατο από τη στιγμή που ε, δεν δίνονται τα απαραίτητα περιθώρια από την κυβέρνηση του Πεκίνου στο Χονγκ Κόνγκ. Όπως σας είπα λοιπόν, εμείς ε, κάναμε και πριν έκκληση για διάλογο, συνεχίζουμε να κάνουμε έκκληση για διάλογο, πιέζουμε τις αρχές του Χονγκ Κόνγκ επ' αυτού και αυτός ήταν και ένας από τους σκοπούς της αποστολής μας την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένης της θέσης του Πεκίνου και του βασικού του ρόλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να θέσει και το θέμα του Χονγκ Κόνγκ κατευθείαν στις αρχές της Κίνας. Ε, πριν είχαμε την ε, αρχή της ε, μίας χώρας δύο συστήματα, αλλά έκτοτε είδαμε ότι οι ίδιες οι αρχές του Πεκίνου έθεσαν το θέμα του Χονγκ Κόνγκ σε μας, ότι έγιναν καταγγελίες, παραπονέθηκαν για εξωτερική ανάμιξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε, να φύγουμε το θέμα με την Κίνα και να επιμείνουμε ότι πρέπει να δώσουν περισσότερα πολιτικά περιθώρια στις αρχές του Χονγκ Κόνγκ για να διευθετηθεί η κατάσταση. Από πλευράς λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, ε, από πείρα ξέρουμε ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία θέση, διότι αν δεν έχουμε, όσο λιγότερο είναι ενιαία η θέση μας ε, κοινή, τόσο λιγότερη είναι η ισχύ μας έναντι της Κίνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τζόσουα. Ελπίζουμε να σε ξαναδούμε σύντομα. Α, θέλεις να προσθέσεις κάτι. Μετά τον νόμο που ψήφισαν ε, οι ΙΠΑ για το Χονγκ η Κίνα ανακοίνωσε κυρώσεις κατά μη κυβερνητικών οργανώσεων, κατά της Human Rights Watch, για παράδειγμα, και μετά την Ιταλική Βουλή, όπου παρέστη ένας βουλευτής της Ιταλίας σε μια ακρόαση, ο πρέσβης του Χονγκ Κόνγκ ε, επέκρινε την στάση του. Πρέπει να πω ότι εγώ ποτέ δεν υποστήριξα ότι θα πρέπει το Hong Kong να είναι ανεξάρτητο. Δεν ε, είμαι ε, υπέρ της απόσχησης. Εγώ ε, θέλω να προωθήσουμε την φιλοδημοκρατική ιδεολογία και την ελευθερία. Καταλαβαίνω ότι η πρόσκλησή σας δεν ήταν κάτι εύκολο διότι υπήρξαν και πολλές επικρίσεις για το Πεκίνο. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση της πάλης μας για την ελευθερία εδώ στο Χονγκ Κόνγκ. Ο κόσμος μας παρατηρεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να θριαμβεύσει η δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόσουα. Γεια σου. Merci <laughs> Περνάμε στο σημείο 4. Η περισσότερη εξωτερική δράση μα έκανε μια δήλωση σε σχέση με το Χονγκ Κονγκ ε, και δεν μπορέσαμε να τη σχολιάσουμε δεν μας δόθηκε ο χρόνος να την σχολιάσουμε. Ο Τζόσου απάντησε. Εσύ λες ότι εμείς δεν απαντήσαμε, έτσι. Η διαδικασία είναι ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, λαμβάνει το λόγο τελευταία πάντοτε μετά τις συζήτησή μας. Οπότε ε, δεν γίνεται συζήτηση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έρχεται να μας ενημερώσει στο τέλος της συζήτησης. Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Έδωσα όμως την ευκαιρία στον Τζόσουα να πει δύο λόγια για να διευκρινίσει μερικά πράγματα. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, καταγγελίες του Πεκίνου ε, ότι πρόκειται για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι υπέρ της απόσχησης. Ε, ε, ήθελε να διευκρινίσει αυτό το θέμα. Δεν νομίζω όμως ότι εμείς μπορούμε να συζητήσουμε την επίσης εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ πρόεδρος ε, δεν πρέπει να μεροληπτεί ε, και, να, και θα πρέπει να είναι ε, ουδέτερη, αλλά ως πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πρέπει να, θέσουμε κάποιο, πρέπει να θέσω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το Βιετνάμ και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Ο κ. Φαν Τσιντούγκ, ε, δημοσιογράφος, ανεξάρτητο δημοσιογράφος, συνελήφθη στις 21 Νοεμβρίου στο Χοτσιμίχ. Το παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου έκανε έκκληση επιγόντω, ε, την οποία δημοσίευσαν και οι New York Times. Ε, ο κ. Ντούγκ έστειλε ένα αίτημα προς τα μέλη του Κοινοβουλίου ζητώντας να αναβληθεί η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ μέχρι ότου λάβουν χώρα σημαντικές βελτιώσεις ε, από την πλευρά της κυβέρνησης του Βιετνάμ. Ο κ. Ντούγκ δεν είναι ο μόνος ο οποίος ε, έχει συλληφθεί. Πολλοί άλλοι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επίσης συλληφθεί επειδή σχολίαζαν την ε, σύναψη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση με το Βιετνάμ. Ήταν μέλη τη κοινωνία των πολιτών που συμμετείχαν στη συζήτηση για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και τη Συμφωνία Επενδύσεων. Εμεί είμαστε Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είμαστε επιτροπή εξωτερικού εμπορίου. Συνεπώ, ο, ο δικό μα ρόλο είναι να γνωμοδοτήσουμε ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο στόχος ε, της νομοδότησης μας αυτής είναι να στείλουμε συγκεκριμένα μηνύματα. Ο κ. Τζόσουα Wong είπε ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε το ρόλο μας. Δεν, έχει καμία, δεν επηρεάζει την κατοπινή συζήτηση, τη μεταγενέστερη συζήτηση, αλλά πρέπει να το πω. Παρακαλώ κύριε Γκέτα. Θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, η πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στην εκτέλεση των καθηκόντων της να, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της, να στείλει μια επιστολή στους πρόεδρους όλων των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου για αυτό για το οποίο μας ενημερώσετε μόλις τώρα. Αυτό θα επέτρεπε εντός της κάθε πολιτικής ομάδας να ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα στο μέτρο που οι πολιτικές ομάδες θα έχουν λάβει μια επίσημη επιστολή από την ε, υποεπιτροπή μας. Πολύ ωραία. Θα στείλω ήδη σήμερα μια επιστολή για το θέμα αυτό σε όλους τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Ο λόγος στην εισηγήτρια Ισαμπέλ Βίσλερ για το θέμα της Συμφωνίας Επενδύσεων και Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών εδώ συμφωνούν, συμφωνεί σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο Βιετνάμ. Και όχι μόνο για την κατάσταση του Βιετνάμ, όσο και για τις δικές μας, τους δικούς μας στόχους, τις δικές μας επιθυμίες. Εδώ υπάρχει μια πραγματική σύγκληση απόψεων. Αν τα πράγματα συνεχίσουν στον δρόμο που κινούνται σήμερα, ε, έχουμε να υποβάλουμε 11 πρωτοβουλίες, 11 προτάσει τροπολογία για την Συμφωνία Εθνών Συναγών και πέντε για τη Συμφωνία Επενδύσεων. Ε, με ξεχωριστή ψηφοφορία. Αυτό δείχνει ε, για το, δείχνει το αποδεικνύει ότι εργαστήκαμε συνενετικά και με αλληλοκατανόηση. Πρόκειται για συμβιβαστικές τροπολογίες και ε, Χαίρομαι που κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά βέβαια και αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες. Μιλήσατε για τους φυλακισμένους του Βιετνάμ. Και εμείς πήραμε πληροφορίες ότι παράλληλα και με λίγο συγκεχημένο τρόπο η... έχει γίνει τροπολογία και της νομοθεσία στο Βιετνάμ και του ποινικού κώδικα αλλά και του εργατικού δικαίου. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να μας στείλουν το μήνυμα ότι το Βιετνάμ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι αντιφατικές οι πληροφορίες, είναι συγκεχημένες. Αυτό δεν είναι πολύ καλό Πρέπει να το πω όμως, διότι πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες έχουν φτάσει στα αυτιά μας τις τελευταίες μέρες. Ελπίζω ότι θα καταλήξουν σε μια συμφωνία α, ικανοποιητική. Το σημαντικό όμως είναι να βελτιώσουμε έστω και ελάχιστα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Ευχαριστώ πολύ όσους συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες. Και τώρα τον ε, λόγο έχει ο κύριος Ραφαέλ Γκλουξμάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η Ιζαμπέλα έδειξε πραγματικά ένα πνεύμα πολύ ανοιχτό, συμβιβαστικό, επιδίωξε τη συνένεση. Και όλοι τελικά έχουμε τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι τελικά αυτό που, σε αυτό που καταλήξαμε είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ δυνατό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως ε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που μένει να καταλήξει. Εάν ε, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, πώς θα ε, εκφράσουμε τελικά, πώς θα διατυπώσουμε το κείμενο. Νομίζω όμως ότι όλοι μαζί ε, θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη μας ότι είμαστε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαιωμάτων και ότι εάν εμείς λοιπόν δεν δίνουμε προτεραιότητα στο, ε, στα δικαιώματα, ποιοι θα το κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα-πρώτα να δώσουμε προτεραιότητα, ε, ναι, στο εργασιακό δίκαιο, ε, οι άλλοι δίνουν προτεραιότητα στο, στην οικονομία. Εμείς όμως θα πρέπει να θέσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πρώτο, στο προσκήνιο. Και αυτή τη στιγμή που εμείς συζητάμε, οι αρχές του Βιετνάμ συλλαμβάνουν άτομα που συμμετέχουν στην διαδικασία διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι έχουμε δίκιο να έχουμε επιφυλάξεις και να θέλουμε να θέσουμε πολύ ισχυρέ προϋποθέσεις πριν υπογράψουμε αυτές τις συμφωνίες. Επομένως, θα συνεχίσουμε να συζητούμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους διότι πραγματικά πολλές φορές ξεκινούσαμε από πολύ διαφορετικές θέσεις, αλλά οι συζητήσεις έγιναν με αγαστή σύμπνοια και ε, αυτό που προέβαλαν οι σοσιαλδημοκράτες εμείς είναι ότι θέλουμε μια πολύ σαφή θέση. Διαφορετικά, το υπόλοιπο Ευρωκοινοβούλιο δεν θα λάβει ξεκάθαρη θέση. Δεν είναι η Ολομέλεια τελικά που θα πρέπει να ε, ε, κυρώσει ή όχι αυτή την συμφωνία. Εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να προβάλλουμε τα δικαιώματα και τη στιγμή που θα καταθέσουμε, ε, που μάλλον προσπαθούμε να διατυπώσουμε αυτή την γνώμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρχές του Βιετνάμ εξακολουθούν να φέρονται με δεσποτικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι σκιώδη εισηγήτρια εδώ και είναι δύσκολο να μιλήσω λοιπόν εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, αλλά συνέβησαν πολλά από την τελευταία μας συζήτηση και θα ήθελα να συζητήσω επομένως για αυτά με την πολιτική μου ομάδα. Χρειάζομαι λοιπόν περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα όμως να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, Ιζαμπέλα, μίλησες για αναθεώρηση του εργατικού δικαίου και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επικρότησε αυτή την αλλαγή, θεωρητικά, αλλά εγώ έλαβα πληροφορίες ότι τελικά αυτή η αναθεώρηση δεν πήγε όσο μακριά θα θέλαμε εμείς. Έχουμε το άρθρο 172 του νέου κώδικα που λέει ότι ε, θα πρέπει όλοι να ανήκουν στην, στις, ε, στον στο, στα εργατικά συνδικάτα του, του Βιετνάμ. Και υπάρχουν και κάποια άλλα άρθρα, τα οποία έχει επισημάνει η Human Rights Watch, το 185, μεταξύ άλλων, στο οποίο θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας. Επίσης, στις 20 Νοεμβρίου ψηφίστηκε αυτός ο νέος νόμος, από ό,τι φαίνεται, και ήταν μία μέρα μετά την ε, σύλληψη του Φανσιντάγκ. Και δεν συλλήφθη μόνο αυτός, αλλά σύμφωνα με τη Human Rights Watch, συνελήφθησαν και 10 άλλοι ακτιβιστές οι οποίοι συνελήφθησαν ή καταδικάστηκαν ανάμεσα στις, την 5η και την 28η Νοεμβρίου. Μετά δηλαδή την επικύρωση του νέου ε, εργατικού δικαίου. Όλα αυτά φαίνονται πολύ ε, αντικρουόμενα. Επομένως, ε, δεν υπάρχουν πολλά που δείχνουν ότι τελικά το Βιετνάμ υποχωρεί στην πίεση που εμείς ασκούμε. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτές τις νέες εξελίξεις και να βρούμε έναν τρόπο για να μπορέσουμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Και έχουμε θέσει κάποιες, κάποιους όρους, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους πριν δώσουμε την έγκρισή μας. Και θα συζητήσουμε στη δική μου πολιτική ομάδα περισσότερο όλα αυτά πριν την επόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ, Ειρήνα κάποιος εκ μέρους των Πρεσίνων. Το ID όχι. Από το ID κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Από το ECR. Κανένας. Από την ΚΟΕ, κανείς. Κανένας λοιπόν από τις πολιτικές ομάδες δεν θέλει να πάρει το λόγο. Ως μέλη. Ως μέλος θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Τζούλη. Um, I'm, not on... Δεν είμαι στην Επιτροπή, στην Αντιπροσωπεία, αλλά ήθελα να ξέρουν τα μέλη ότι έχω, κανονίσει, έχω οργανώσει μία συνάντηση αύριο με ανθρωπιστικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να μιλήσουμε για την περιπλοκότητα αυτού του θέματος, αυτής της ασυνέπειας που υπάρχει, της αντίφασης που υπάρχει. Θα πρέπει να έχετε λάβει προσκλήσεις για την εκδήλωση αυτή. Αν σας ενδιαφέρει να έρθετε, πραγματικά θα ήθελα την, εμπειρία σας, γιατί εσείς ασχολείστε άμεσα με το θέμα αυτό, ενώ εγώ απλώς ε, απάντησα στο, στην έκκληση ε, των ε, οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν να... Ε, είναι πολύ χρήσιμο για μένα που είμαι τώρα εδώ για να δω πώς ακριβώς διαχειρίζεστε εσείς το θέμα. Μισό λεπτό να βρω και τι ώρα είναι η συνάντηση αύριο. Αύριο... Στις, από τις 12 ως τις 2 στο ASP G315. Ε, μπορεί να μάθει και εσείς κάτι καινούριο από τις οργανώσεις αυτές με τις οποίες θα μιλήσουμε. Οπότε, ελάτε παρακαλώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο για το φάκελο για το Βιετνάμ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Ε, επειδή δεν μίλησε κανένας από τη δική μου την ομάδα. Να πω ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ του να δοθεί συνένεση στη συμφωνία με το Βιετνάμ, για την εμπορική αυτή συμφωνία, κυρίως όταν επιβάλλουν μέτρα καταστολής σε ανθρώπους που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχουμε δει. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να πιέσουμε λίγο, να επιμείνουμε το Βιετνάμ να μας ξεκαθαρίσει λιγάκι διάφορα θέματα που του έχουμε θέσει πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για ολοκλήρωση των εμπορικών αυτών συμφωνιών και συναλλαγών. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα την υπηρεσία των εξωτερικών δράσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμάς μας ανησυχούν οι τελευταίες ε, συλλήψεις που έχουν καταγραφεί. Το έχουμε θέσει και μέσω της επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας και στο το δυνατό επίπεδο στο Βιετνάμ, εκφράζοντας την ανησυχία μας. Έχουμε μια σχέση που εξελίσσεται γενικώ με το Βιετνάμ επί τη βάση διαφόρων συμφωνιών που έχουμε κάνει και αποτελούν την ε, προετοιμασία και για την εφαρμογή και στα πλαίσια του IPA και των ε, ανθρωπίνων ε, ε, των εμπορικών συμφωνιών. Έχουμε την ε, συμφωνία FLECT για το ξύλο, έχουμε τη συμφωνία της 25ης Οκτωβρίου, όπου το Βιετνάμ μπορεί να πηγαίνει στις υπηρεσίες, να παίρνει μέρος μάλλον στις αποστολές άμυνας. Έχουμε λοιπόν διάφορων, διάφορων ειδών συμφωνίες και έχουμε αρκετά θετικές εμπειρίες από τη συνεργασία με το Βιετνάμ και στο ΑΣΕΑΝ και βεβαίως Περιμένουμε το 2020 στο Βιετνάμ να αναλάβει και την Προεδρία του, Ασια, του ΑΣΕΑΝ. Η PCA είναι το πλαίσιο βάθυνση των ε, σχέσεών μας και μέσω αυτού το Βιετνάμ έχει δεσμευθεί να σέβεται τις αρχές ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές ε, καταγράφονται και στα ε, μέσω των διακήρυξεων των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν υπάρξει, έχει υπάρξει πρόοδος ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο ρυθμός φτώχειας έχει μειωθεί δραματικά και ως αποτέλεσμα αυτής της πρόοδου έχουμε δει και κάποιες σημαντικές εξελίξεις και στα οικονομικο-κοινωνικά δικαιώματα, αλλά βεβαίως φυσικά συμμεριζόμαστε τις ανησυχίε του Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και την κατάσταση ε, των ε, ε, υπεραμεινόμενων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συστηματικά θέτουμε τα θέματα αυτά στις αρχές, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο στο Βιετνάμ και ε, συχνά το θέμα αυτό των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπαίνει ως σημείο συζήτησης στον διάλογο, στο σχετικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου συζητούμε επιμέρους υποθέσεις. Ο διάλογος αυτός είναι όντως μια αργή διαδικασία, αλλά έχει δώσει αποτελέσματα σε κάποιους τομείς. Οι συζητήσεις αυτές δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά ο διάλογος πάντα λαμβάνεται στα σοβαρά από τους ε, α, Βιετναμέζους και βεβαίως πάντα μπαίνουν όλα τα θέματα στο τραπέζι των συζητήσεων και σίγουρα τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση σε σχέση με την αφοσίωση που δείχνει το Βιετνάμ σε αυτά τα θέματα, σε σχέση με το που ήμασταν πριν από λίγα χρόνια. Ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίση έχει βοηθήσει και την ε, αντιπροσωπεία στο Ανόη ε, να προωθήσει το θέμα των ε, υπεραμεινωμένων, των ακτιβιστών μέσω τριμερών διαλόγων, πρόσβαση στο νομικό συμβούλιο κτλ. Οπότε προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε το Βιετνάμ στο θέμα αυτό, στις συζητήσεις και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε είναι σημαντικό να έχουμε την IPA αλλά και την FTA, την ε, Συμφωνία για το ε, Ελεύθερο Εμπόριο. Αυτές οι, σημασίες, αυτές οι συμφωνίες συγγνώμη, θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά με το Βιετνάμ. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και ευχαριστώ. Θέλει η Κομισιόν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. από τη Γενική Διεύθυνση Trade ε, είμαι. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω. Να πω κάτι που είπατε κι εσείς, κυρίως στο θέμα του χρονισμού. Όλοι νομίζω συνειδητοποιούμε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή η συμφωνία. Αλλά ας μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε. Εγώ έχω εμπλακεί σε όλες τις συμφωνίε ε, ελεύθερου εμπορίου, σε όλα τα κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη και αν σκεφτώ κάποιου άλλου τέρους, ε, το Βιετνάμ έχει πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Πριν από δύο χρόνια δεν υπήρχε τίποτα για τη μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου. Είχαμε δύο ε, εκπροσώπους από τη Μολύσα που προσπαθούσαν να προωθήσουν μια αλλαγή. Αν δούμε τώρα που έχει φτάσει το πράγμα, έχουν ε, τον νέο εργασιακό κώδικα, έχουμε την επικύρωση της νομοθεσίας του 98, έχουμε έναν οδικό χάρτη για την ε, διακήρυξη 87 ε, και 105, Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για του χρόνου, όπου ξεκινούν να δουλεύουν για, στα σχέδια εφαρμογής. Ξέρουν ότι πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία για τα συνδικάτα. Οπότε, εντάξει, είναι τέλειο. Όχι, είναι το, ε, το ποτήρι γεμάτο. Όχι, είναι μισό γεμάτο όμως. Αν δεν μπούμε τώρα στην διαδικασία αυτή, τι θα γίνει είναι σαφές ότι εκτός του Βιετνάμ υπάρχουν και στενοί εταίροι του Βιετνάμ, ένας πολύ μεγάλος μάλιστα, που δεν του αρέσουν και ιδιαίτερα αυτές οι μεγάλες αλλαγές. Έχει αρκετή πίεση λοιπόν το Βιετνάμ να μην συνεχίσει αυτές τις ε, εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Οπότε είναι πραγματικά μεγάλη η αφοσίωση του Βιετνάμ στις συμφωνίες αυτές. Έχουμε εδώ και δύο χρόνια ξεκινήσει, αλλά τώρα είναι πολύ εντατικοποιημένες οι προσπάθειες. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε αποστολή, οπότε τώρα πρέπει να κλειδώσουμε όλα αυτά τα σημεία, όλα αυτά τα βήματα, έτσι ώστε το σχέδιο μάχης ε, να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί τελικώς η συμφωνία. Και να προσθέσω Νομίζω ότι οι συνάδελφοί σας στην ε, Επιτροπή τα πρόσφατα πήγανε στο ε, Βιετνάμ και είπανε ότι είναι καλή, ακόμη και οι ντόπιοι, ακόμη και οι ε, μπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία στο Βιετνάμ λένε ότι είναι καλύτερο να έχουμε αυτή τη συμφωνία. Ε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς να κινητοποιηθούμε καλύτερα και μιλούμε για μια κυβέρνηση που έχει δεσμευθεί να ε, εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή. Οπότε τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία γιατί αλλιώ σε δύο-τρία χρόνια δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν βεβαίω υπάρχουν ερωτήσει ή τεχνικά σχόλια που θέλετε να απαντήσω, εδώ είμαι. Merci. Je vais respecter la règle θα σεβαστώ τον κανόνα να μην σας δώσω το λόγο. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε άπειρα πράγματα σε σχέση με αυτά που είπατε. Δεν έχουμε χρόνο όμως. Νάτσο. Ε, απευθύνομαι σε σένα και σε όλους τους αδέλφους της Επιτροπής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ακρόαση με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων κάποια στιγμή για αυτό το θέμα. Τώρα δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Για να γίνει κάτι τέτοιο, λέει η Πρόεδρο, υπάρχει μία λύση. Την Τετάρτη, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η ΑΦΕΤ, να ψηφίσει την αναβολή. Σε αυτή την περίπτωση θα συζητήσουμε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, να κάνουμε, να διοργανώσουμε ακροάσεις πιο σημαντικές. Γιατί θα μπορούσαμε να δούμε το ποτήρι ως μισοάδιο ή ως μισογεμάτο. Αυτό είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε πάντως σίγουρα να το γεμίσουμε περισσότερο και χρειάζομαστε χρόνο γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες συμφωνίες οι οποίες περίμεναν χρόνια και χρόνια πριν εγκριθούν. Γιατί για να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο απαιτήσεων ως κοινοβούλιο. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο για την συμφωνία με το Βιετνάμ. Θα δώσω το λόγο στην Ισαμπελ Βίσλερ που είναι η συγγήτρια που ενδεχομένω θα προτείνει την ε, αναβολή η ίδια όμως θα κάνει την πρόταση αν το αποφασίσει. Δεν είχα την ε, πρόθεση να μιλήσω ούτε για συνένεση, συγκατάσταση, ούτε για απόρριψη, ούτε για αναβολή. Γιατί ε, έχει γίνει μόνο μία τυπή συνεδρίαση μέχρι τώρα μεταξύ μας και δεδομένου ότι <laughs> έγινε αυτή η μικρή συζήτηση μετά την παρέμβαση Κομισιόν, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις ε, ανάλογα με τις πεπιθήσεις του καθενός. Όλοι, θέλουμε τον, ε, όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο όλοι έχουν τον ίδιο στόχο. Ο καθένας ε, δίνει λόγο στη συνείδησή του ε, και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το ποιο θα πρέπει να είναι ο δρόμος για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε να ζητήσουμε αναβολή. Προτάθηκε αυτό, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει συνένεση αυτή η πρόταση. Υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ λύσει και άλλε δυνατότητε που θα μα επέτρεπαν να ακολουθήσουμε αυτή την, την άγουσα που θα μας επιτρέψει να έχουμε ίση τη, τη συνείδησή μας. Ο κ. Γκέτα, για να βοηθήσω τη συζήτηση, όχι για να απαντήσω στην Κομισιόν. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να συμφωνήσουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή ότι αυτή, τούτη εδώ η Επιτροπή θα πάρει μια θέση υπέρ, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, την αναβολή, υπέρ της αναβολής, υπέρ της αναστολής, υπέρ της πιο ε, λεπτομερούς ανάλυσης, ίσως αυτό, ε, σε, σε περισσότερο βάθος, ανάλυση σε περισσότερο βάθος, ίσως αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, του θέματος. Αν μπορούσαμε δηλαδή να συμφωνήσουμε σε αυτή την ιδέα μια, υπέρ μια πιο λεπτομερού εξέτασης ή ανάλυσης της συμφωνίας. Ίσως αυτό ε, θα ε, έδινε κάποιο, κάποια ευκαιρία στις υπόλοιπε επιτροπές και στις πολιτικέ ομάδες να προβληματιστούν και να δούμε το αποτέλεσμα. Ο ρόλος μας πάντως ε, είναι να είμαστε ε, αυτοί που θα σημάνουν συναγερμό, αυτοί που θα εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη φροντίδα για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Γκλουξμαν. Ε, συμφωνώ με την Ισαμπέλ, η συζήτηση ακόμα διεξάγεται, δεν έχει ολοκληρωθεί μεταξύ μας, οπότε ίσως ε, θα μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο να δείξουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμα από τις τελευταίες εξελίξεις. Εγώ όμως έχω μια ερώτηση προς την Πρόεδρο. Είναι λίγο ε, πιεστικός ο κανόνα αυτό να μην μπορούμε να πάρουμε το λόγο μετά την Κομισιόν. Πώ θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε αυτόν τον κανόνα. Ε, θα, το συζητήσουμε στο, θα το συζητήσουμε στη συνεδρία τη συντονιστών. Η... Ζητήθηκε η γνωμοδότησή μας για, αυτές τις δύο... για αυτά τα δύο κύματα. Η γνώμη της υποεπιτροπής μας ε... ε πρώτον αφορά τη συγκατάθεση όχι. Οπότε εκεί δεν προδικάζω το αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τρία πράγματα. Ή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας, οπότε συμφωνούμε με την επενδυτική συμφωνία, είτε την απορρίπτουμε και τις δύο συμφωνίες, έτσι μιλώ και για τις δύο συμφωνίες, ε, ή αναβάλουμε. Ναι, όχι ή αναβολή. Τρία πράγματα, τρεις είναι οι επιλογές. Δεν έχουμε κάποια τέταρτη. Σε αυτή τη θέση μας, σε αυτή την απόφασή μας, όταν ληφθεί, μπορούμε να συνάψουμε, να επισυνάψουμε και ένα ψήφισμα. Συνοδευτικό. Όπως ε, είπε και η συγγήτρια, υπάρχει μια σημαντική σύγκληση απόψεων σε σχέση με αυτό το ψήφισμα. Όμως το σημαντικό είναι η πρώτη μας φορία υπέρ, κατά ή αναβολή. Αν δεν συμφωνήσουμε σε μία από αυτέ τι τρει επιλογέ δεν μπορούμε να επισυνάψουμε και κανένα ψήφισμα. Αυτοί είναι οι κανόνε. Καλή, κακή, δεν έχει σημασία. Και με βάση αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να εργαστούν οι εισηγήτρια και οι συνεισηγητές. Έτσι ώστε την Τετάρτη να λάβει χώρα η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Όχι εδώ, η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό είπα στον Νάτσο προηγουμένω. Αν θέλουμε να παρατείνουμε να επιμηκύνουμε τη συζήτηση, δεν μπορεί να γίνει αν δεν αναβληθεί η ψηφοφορία τη ΑΦΕΤ. Εμεί θα πρέπει να υποβάλουμε την γνωμοδότησή μα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Ε, και θα ήταν κρίμα να μην πάρουμε, να μην εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να εκφέρουμε γνώμη για μια συμφωνία η οποία αφορά την ε, σοσιαλιστική κομμουνιστική δημοκρατία του Βιετνάμ που είναι και αυταρχική σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κρίμα θα ήταν. Αλλά μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει μέχρι Τετάρτη. Δηλαδή, παρά τη συνένεση των πολιτικών ομάδων, ενδεχομένως το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να μην εκφέρει γνώμη για τις συμφωνίες αυτές με το Βιετνάμ. Μπορεί, είναι δυνατόν. Θα αφήσω όμως το θέμα αυτό στα χέρια της εισηγήτρες και των σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω να μην καταλήξουμε σε τέτοια ε, κατάσταση. Δηλαδή, η, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ζήτησε να γνωμοδοτήσει, να μην γνωμοδοτήσει τελικά. Ειρήνα, νομίζω ότι με κάλυψες. Πρόεδρος. Ωραία, κλείνουμε το θέμα. Αφήνω το θέμα στο την εισηγήτρια και του και εισηγητέ, προκειμένου να καταλήξουμε στην ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Τετάρτη. Κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν περάσουμε στο σημείο 8 σε λίγο.